liebe Kolleginnen und συνάδελφοι, με 40 λεπτά καθυστέρηση ξεκινάμε την ε, συνεδρίασή μα. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που έπρεπε να περιμένετε, αλλά οι, οι κοινέ ψηφοφορίε με την Επιτροπή απασχόληση ε, πήραν λίγο παραπάνω από ό,τι είχαμε υπολογίσει, οπότε πραγματικά ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Πριν ξεκινήσουμε και δούμε την ακρόαση, να πω ότι σήμερα το πρωί είχα πει, είχα ανακοινώσει ότι θα ε, απέσυρα το όνομά μου από τον ε, ε, σχετικό κανονισμό. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση. Οι συνάδελφοι κατάλαβαν ότι το έχω ήδη κάνει. Όχι, δεν το έχω κάνει, απλώς είπα ότι θα το κάνω, θα το εξέτασα κτλ. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη, θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν, ε, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ήθελα, οπότε... αποφάσισα τελικά να προσπαθήσω να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα της Επιτροπής μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε τώρα στην ακρόαση. Στις ε, 20 Ιουνίου πριν ε, περίπου ένα χρόνο, 2016, ε, έγινε, η, έγινε το δημοψήφισμα για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 51,9% των Βρετανών ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης. Στις 21 Μαρτίου 2017 η Ηνωμένη, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε την ε, αίτησή του για την αποχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη την ώρα λοιπόν, εκείνη την ημέρα ξεκίνησε να, να κυλάει ο χρόνος για την ε, περίοδο των δύο ετών των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, ξεκίνησαν λοιπόν οι διαπραγματεύσει την ε, ε, Δευτέρα. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα σε σχέση με το μέλλον, νομίζω ότι ακόμα είμαστε όλοι σε μία ομίχλη. Οι πολιτικές συνθήκες που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αλλάξει από τότε που η ε, Πρωθυπουργός ε, έστειλε το αίτημά της για την αποχώρηση θα δούμε τώρα ποιε θα είναι οι νέε νέες σχετισμοί δυνάμεων στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα προς το παρόν δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Πρέπει να περιμένουμε. Στην Επιτροπή Πολιτισμού ελπίζουμε ότι και τις, για τι δύο πλευρές αυτές οι διαπραγματεύσει θα έχουν τελικά ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος γιατί ουσιαστικά μιλούμε για, την, για τα συμφέροντα των πολιτών μας αλλά και, για, και, και των ε, τωρινών πολιτών μας και για, τον, για του μελλοντικού πρώην πολίτε μας του Βρετανού πολίτε δηλαδή δηλαδή. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ εδώ στην Επιτροπή μας και ε, με μεγάλη πλειοψηφία καταψήφισαν το Brexit. Και κυρίω και αυτό με τους ε, φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και όλες τις επιχειρήσεις ε, που βρίσκονται στον δημιουργικό τομέα και που διαστηριοποιούνται στην Ευρώπη των 27 αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τους ε, σημερινούς λοιπόν υπερογνώμονές μας θέλουμε να ασχοληθούμε με την ακρόαση αυτή και με τη βοήθειά τους να δούμε ε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο, στο μέλλον. Να δούμε δηλαδή ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit και για τους Βρετανούς αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ποιες είναι οι εταιρικέ σχέσεις που θα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Γι' αυτό έχουμε πέντε εμπειρογνώμονες σήμερα από τον ακαδημαϊκό τομέα. Έχουμε, ε, τους έχουμε καλέσει στην Επιτροπή μας, για, θα τους παρουσιάσω και βεβαίως τους ευχαριστώ ήδη για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Και πάλι ζητώ και από αυτούς συγγνώμη που ξεκινούμε τόσο αργά. Να πω ότι πραγματικά λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν παρίσταται σήμερα. Δυστυχώς ο ε, ε, επικεφαλής διαπραγματευτής, ο κύριος Μπαρνιέ, δεν μπορούσε να δεχτεί την πρόσκλησή μας λόγω του φόρτου εργασίας, κατανοητό βεβαίως αυτό. Βεβαίως και ο ο Γκίφερ Χόφστατ που είναι ο δικό μα εκ, εκ μέρου του Κοινοβουλίου επικεφαλή διαπραγματευτή δεν μπορούσε να δεχτεί την πρότασή μα να είναι παρόν σήμερα εδώ. Είναι κρίμα, αλλά νομίζω ότι α, κατά τη διάρκεια τη ε, όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα έχουμε αρκετέ ευκαιρίε να συνδιαλλαγούμε μαζί του. Και επίση ε, η Γενική Διεύθυνση για την ε, εκπαίδευση και τον πολιτισμό δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και αυτό είναι λυπηρό θα χρειαζόμασταν την υπερογνωμοσύνη τους, θα μας βοηθούσε, αλλά δυστυχώς και αυτό δεν ήταν δυνατό. Παρ' όλα αυτά, η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης μας έστειλε γραπτός κάποια α, σημαντικά στοιχεία, ε, σχόλια, αριθμητικά στοιχεία κτλ. Υπάρχουν όλα στους φακέλους σας. Σε τρία μικρά πάνελ έχουμε χωρίσει τη σημερινή ακρόαση. Κάθε εμπειρογνώμων θα μιλήσει για το πολύ 10 λεπτά και μετά από αυτά τα πάνελ θα έχουμε μία σύντομη α, περίοδο ερωτήσεων και απαντήσεων. Βεβαίως πρέπει να είναι λίγο το πιο αυστηρό το χρονοδιάγραμμά μας γιατί ε, καθυστερήσαμε. Να ευχαριστήσω και, την, ε, και τα μέλη. Βεβαίως θα σας δώσουμε τον ε, χρόνο να μιλήσετε, να παρέμβετε, να θέσετε ερωτήματα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε καταρχάς τους ομιλητές του πρώτου πάνελ, ο κύριος, ο καθηγητής Τζαντονάτο Κατζάνο. Ελπίζω να το, προ, να το προέφερα σωστά. Ε, είναι καθηγητής νομικής στην ε, Ρώμη και επίσης είναι ο εκδότης της, ε, του νομικού περιοδικού Studi sull'integrazione europea. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε αυτό. Ε, θα μας παρουσιάσει ποιες είναι οι μορφές εταιρικών σχέσεων που θα, μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Μεγάλης Βρετανίας. Κύριε Κατζάνο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής επί ενός θέματος το οποίο είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικό και βεβαίως ε, επίκαιρο και για τους νέους αλλά και για το μέλλον του πολιτισμού, καθώς επίσης και το μέλλον των πανεπιστημίων, αλλά και όλων όσοι ασχολούνται με την δημιουργία. Ε, αναφερόμαστε λοιπόν σε ε, μια μεγάλη ενεργητικότητα για την Ευρώπη. Ε, αυτή η μεγάλη ενέργεια η οποία ε, δημιουργεί οικοδομή αυτήν την Ευρώπη η οποία είναι ισχυρή, ε, δύναμη κατά την έννοια αυτή σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι μπορεί κανείς να έχει την αίσθηση ότι το θέμα της εκπαίδευσης ε, ε, είναι και του πολιτισμού είναι ένα εύκολο στοιχείο στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, διότι στις συνθήκες δεν υπάρχει πρόβλεψη εναρμόνισης νομοθετικής για, αυτό, για αυτή την αρμοδιότητα, όπως ε, συμβαίνει στις άλλες ε, που είναι μικτές ή αποκλειστικές αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει επομένως ε, νομοθεσία και άρα οι οδηγίες και οι κανονισμοί που έχουν εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν θα πρέπει να έχουν ε, τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην περίπτωση του Brexit. Αυτό όμως είναι εσφαλμένο ως θέση, διότι στην πραγματικότητα ο πολιτισμός και η εκπαίδευση πέρα από τα σημαντικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν και θα αναφέρω μάλιστα σε λίγο, σημαντικά ε, προγράμματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και πολιτιστικής δημιουργίας, πέρα από αυτά λέω υπάρχει και μία σειρά ε, ευνοσιακής νομοθεσίας ε, που έχουν μειωμένη εδαφική μειωμένο δαφικό αντίκτυπο. Ας πούμε, η επιστροφή π.χ. πολιτιστικών αγαθών από την επικράτεια ενός κράτους μέλους, εναρμόνιση των ε, νομοθεσιών όσον αφορά ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, ή επίσης όλες οι προϋποθέσεις εργασίας στην βιομηχανία του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Η πολιτιστική διάσταση επίσης στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδήποτε και η αναγνώριση των διπλωμάτων που είναι ένας άλλος τομέας σημαντικός και η ελευθερία εγκατάστασης ε, των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών Ινστιτούτων από τη μία χώρα στην άλλη και βεβαίως ε, ε, τελευταίο και πολύ σημαντικό η κυκλοφορία των φοιτητών αλλά και των καθηγητών. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να συζητηθούν διότι θα φυγούν από αυτήν την δραματική περίσταση του Brexit που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Όλο η δέσμη ε, αφορά το κεφάλαιο 26 ε, όπως ας πούμε βλέπουμε και στις διαπραγματεύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και με τη Σερβία. Υπάρχει εκεί ένα κεφάλαιο 26 το οποίο αναφέρεται ε, στην, στο κεκτημένο για την εκπαίδευση και για τον πολιτισμό και αρκεί κανείς να δει αυτά τα δύο παραδείγματα της Σερβίας δηλαδή και της Τουρκίας για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Επομένως αυτή η διαδικασία η οποία ξεκινάει τώρα που ξεκίνησε μάλλον χτες, είναι μία διαπραγμάτευση η οποία αφορά το διαζύγιο, την απόσυρση, αλλά μήπως ταυτόχρονα είναι και η διαπραγμάτευση για μία ή περισσότερες συμφωνίες που θα αφορούν το μέλλον των σχέσεων. Αυτό ακόμα σήμερα ε, δεν ε, λαμβάνει ίδια απάντηση. Και, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση δεν είναι ίδια από πλευράς της Κομισιόν και από πλευράς Λευκής Ευήβλου ε, και Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα διαπραγματευόμαστε ας πούμε δύο ε, συμφωνίες, δύο ομάδες συμφωνιών ή μονάχα την απόσυρση. Εγώ νομίζω ότι πιο πιθανό είναι το δεύτερο σενάριο, δηλαδή της αποχώρησης ε, το οποίο μετά θα ακολουθήσει ε, και η διαπραγμάτευση επί μιας ή περισσότερων συμφωνιών που θα αφορούν το μέλλον. Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον. Πολλές ε, είναι οι απόψεις και πολλά μοντέλα έχουν μελετηθεί και όλοι εσείς άλλωστε φαντάζομαι ότι έχετε κάποια αίσθηση των πολλών πιθανών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, αυτά τα μοντέλα ας πούμε, ή το πιο γενικό ε, μοντέλο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ε, ή επίσης το μοντέλο της, ε, του Καναδά βάσει της Εμπορικής Συμφωνίας με τον Καναδά. Θα πρέπει να, να δει κανεί βέβαια και το περιεχόμενο όλων αυτών των μοντέλων, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχουν λειτουργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προβλέπουν ε, κάποια στοιχεία εμπορίου, προβλέπουν κάποια στοιχεία ε, ε, ελεύθερη κυκλοφορίας ατόμων που αποτελεί μία από τις τέσσερι ελευθερίε. Θα ήθελα να πω στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου ότι η συμφωνία με την Τουρκία παρουσιάζει ε, μία σημαντική ιδιαιτερότητα ε, που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αξιολογήσει ε, και συμπεριλάβει σε πολλές αποφάσεις. Όταν εγκρίθηκε η απόφαση 180 της Συμφωνίας Σύνδεσης εισήχθη στι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, που τότε ήταν ακόμα Ευρωπαϊκή Κοινότητα και της Τουρκία, εισήχθη λέω ε, η λεγόμενη Stand Still Clause μία ρήτρα λοιπόν ε, η οποία έλεγε ότι δεν θα μπορούσε ε, να τροποποιηθεί πλέον η θέση με συσταλτική ερμηνεία η θέση των Ευρωπαίων εργαζομένων στην Τουρκία και των Τούρκων εργαζομένων την Ευρώπη. Πολλές ε, ε, δικαστικές αποφάσεις είχαμε. Ε, εγώ αναφέρω μονάχα τη Συμφωνία Ντερέτσι, στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέφερε ότι από την συμφωνία με την Τουρκία μπορούσαν να βρεθούν ε, κάποια στοιχεία τα οποία μπορούσαν ε, να αντιταχθούν κατά κάποιο τρόπο στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, βεβαίως, το εμπαρόδο ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα δύο στοιχεία να συγκριθούν. Από την άλλη πλευρά ε, αναφερόμαστε ε, ε, στην ουσία αν και κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία του 2004 που προβλέπει η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και της οικογένειάς τους. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή αναφορά σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία αφορούν την ακρόασή μας. Επομένως, έχουμε τους δύο μεγάλους τομείς το, της εκπαίδευσης, education, των, ε, ε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακών σπουδών κτλ. Και έχουμε από την άλλη μεριά τον τομέα της δημιουργίας ε, ε, και της δημιουργικότητας. Στον έρασμο, ας πούμε, μπορεί κανείς να πει ότι τελικά είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια διότι οι γενναίες, των, ε, ε, ε, οι νέοι άνθρωποι μάλλον, η νέα γενιά μπορούσε να έρθει σε επαφή. Μάλιστα πρόσφατα γιορτάσαμε και την, το, γενέθλιο αυτό, την επέτειο των 30 χρόνων του Εράσμους, που είχε πραγματικά πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί αυτή η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δέχεται πάρα πολλές αιτήσει από τους τους ε, νέους των 27 άλλων χωρών ότι δεν θα συμμετάσχει πλέον. Ποιο είναι όμως το κεντρικό ερώτημα. Το κεντρικό ερώτημα είναι και λυπούμε που το λέω αλλά μπαίνουν ε, ε, και οικονομικά στοιχεία. Το ζήτημα λοιπόν είναι το λεγόμενο entry ticket για να συμμετάσχει μία χώρα για να μπορέσει να συμμετάσχει μια χώρα. Στο Εράσμου θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική υπηρεσία και θα πρέπει να ε, ε, πληρώσει και κάποια χρήματα, γιατί έτσι δεν θα πληρώνουν τα παιδιά, δεν θα πληρώσουν δηλαδή τους ε, τα... τη συνδρομή εγγραφής και θα πάρουν μια υποτροφία. Το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως θα μπορούσε να φυγεί και να γίνει τρίτη χώρα διότι το έρασμος προβλέπει και την συνεργασία τρίτων χωρών. Ε, και η Τουρκία επίσης ε, συμπεριλαμβάνεται όπως και άλλες χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα μπορούσε να διαφοροποιείται αναπερίπτωση. Ξέρετε ότι υπάρχουν κατηγορίες προγραμμάτων Εράσμους που είναι τέσσερις αλλά η, συνολική δέσμη, το συνολικό πακέτο προβλέπει την πλήρη συμμετοχή, full partnership αυτό το πακέτο θα πρέπει να το διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα άλλο παράδειγμα, ένα άλλο μοντέλο είναι το μοντέλο της Ελβετίας. Το 2014 ε, ε, η Ελβετία συγγνώμη, καταψήφισε την ελεύθερη κυκλοφορία των φοιτητών και εκεί υπήρξε μια μεγάλη δυσκολία. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί ε, η κυκλοφορία μέσω έρασμους είναι ελεύθερη κυκλοφορία ή μπορεί να υπάρξουν και κάποιες εναλλακτικές. Αυτό συνέβη στην ε, Ελβετία και είναι αρκετά ενδεικτικό. Στην ουσία λοιπόν η συμμετοχή της Ελβετίας πάγωσε και όχι για λόγους τιμωρητικούς απέναντι στην Ελβετία, ε, διότι οι πολιτικοί δεσμοί ε, και οι νομικοί δεσμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ε, να αναφέρω την σχέση ανάμεσα στο ε, Europass και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, γιατί νομίζω ότι το ένα έχει νομικό χαρακτήρα, το άλλο έχει και, και επομένως δεσμευτικό, το άλλο έχει εθελοντική βάση. τα γνωρίζετε αυτά νομίζω ότι είναι κρίμα να μην σκεφτούμε λίγο και το θέμα ε, των ε, ε, όλων των έργων της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου κτλ. Πολύ πρόσφατα, τον Απρίλιο μάλιστα, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο η ενιωστή, η μάλλον ε, μεταρρύθμιση ε, της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς ε, σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο οπτικοακουστικός τομέας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Υπάρχουν πλατφόρμες πλέον οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον έτσι ώστε να δει κανείς έργα, φιλμ, ταινίες είτε για να ακούσει μουσική και επομένως εάν το Ηνωμένο Βασίλειο βγει από αυτήν την διαδικασία τότε αυτό θα αποτελέσει πραγματικό ακροτηριασμό του οπτικοακουστικού ε, τομέα ε, και ε, κατανοούμε νομίζω όλοι ότι ένας οπτικοακουστικός τομέας με πλατφόρμες οι οποίες δεν θα έχουν και τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν πραγματικά κάτι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και πάλι συγγνώμη που σας πιέζω λιγάκι, αλλά ε, για να είμαστε δίκαιοι και με τους ε, υπόλοιπους προσεκλημένους, να έχουν χρόνο και αυτοί να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να χαιρετήσω 14 φοιτητέ και φοιτήτριε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Καλή ημέρα διαλέξατε για να έρθετε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα σας ενδιαφέρει πολύ το Brexit. Οπότε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Δρογεύσκη έχει πρώτος το λόγο. πρόεδρο, πρόεδρος της μικρής εποπτικής ομάδας για το Brexit από την Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο ένα λεπτό μόνο, γιατί μέχρι τις 5 ε, και 4 πρέπει να τελειώσουμε για να συνεχίσουμε. Przykłady wymienione przez Pana są interesujące, natomiast e, ta lista będzie rzeczywiście... Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αν μιλάμε τώρα για ε, έργα τέχνης και τα λοιπά, έχουμε, είναι πάρα πολλές ε, οι ανταλλαγές που υπάρχουν, έχουμε πάρα πολλά έργα τέχνης τα οποία βρίσκονται σε μουσεία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Φυσικά είναι και πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ερευνητών που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ε, είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος όλων αυτών των ανταλλαγών που έχουμε. Θα ήθελα να μου πείτε από πότε και μετά ε, θεωρείτε ότι μπορεί να αρχίσει η καταγραφή ε, όλων αυτών των έργων κτλ. Ε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια ε, έγγραφα τα οποία είναι, δεν είναι ακριβώς δημόσιας πρόσβασης και επομένως θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Επίσης, ακόμα και στον τομέα του τουρισμού μπορεί να υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι απόρριτα και τα οποία στα οποία δεν θα έχουν πρόσβαση όλοι. Τι γίνεται με αυτά. τελευταία παρατήρηση για τους φοιτητές έχοντας ως δεδομένο ότι από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2019 ξαφνικά ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα νομικό κενό. Γιατί μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχουν φοιτητέ οι οποίες βρίσκονται ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανοί οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ευρώπη. Τι γίνεται με αυτούς. Ευχαριστώ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Κατζάνο. Καταλαβαίνω ότι τα 10 λεπτά ε, είναι πραγματικά πολύ λίγα και πάρα πολύ δύσκολο να κάνει εξαντλητική παρουσίαση σε τόσο μικρό ε, χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όλα αυτά, δώσατε κάποιες ε, οδούς σκέψεις. Αναφερθήκατε στο μοντέλο της Νορβηγίας, της Ελβετίας. Αναφερθήκατε στο μοντέλο σχέσης σαν αυτό που έχουμε με την Τουρκία. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτούς διάβλους ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και με όλους τους υπόλοιπους λαούς, ε, όσον αφορά την δημιουργία και την εκπαίδευση. Αλλά μία από τις προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να συμμετάσχει στο Εράσμους είναι ακριβώς να σέβεται την αρχή της κυκλοφορίας των ατόμων, αλλά βεβαίως και να συμμερίζεται κοινέ ε, ε, αξιακές αρχές, καθώς επίσης φυσικά ε, να πληρώνει και την οικονομική συμβολή αν ε, ε, ε, απομακρυνθούμε από το hard Brexit και καταλήξουμε σε μία λύση τύπου ελευθέρου οικονομικού χώρου, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε πιο εύκολα μία λύση αλλά νορβηγικά. Εάν όμως ε, ε, φτάσουμε στο hard, στο σκληρό Brexit, στο ακραίο Brexit, τότε οπωσδήποτε το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ε, σαν, την, σαν μια οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν τρίτες χώρες ε, οι οποίες ε, συμμετέχουν σε προγράμματα όπως ας πούμε Δημιουργική Ευρώπη, αλλά ε, θα πρέπει ως προϋπόθεση να ενστερνίζονται την οδηγία. Δηλαδή για να αντιστρέψω το σκεπτικό δεν είναι ότι αποκλείει η οδηγία, είναι ότι εάν Εάν ε, ε, η χώρα δεν βρίσκεται μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενστερνίζεται την οδηγία. Ε, αυτά ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Julie Ward. I think... Νομίζω ότι αναγνωρίσατε ένα από τα βασικότερα προβλήματα όταν χρησιμοποιήσατε τη λέξη ενέργεια. Η ενέργεια, η δημιουργία και το πάθος που προέρχεται από την ευκαιρία του να ε, ζήσει κανείς και να φοιτήσει σε μια άλλη χώρα ώστε να μπορέσει να ερωτευτεί έναν άλλο τρόπο ζωής ε, είναι ένα από τα ε, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του Brexit τα δικαιώματα των παιδιών επίση είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα θεωρούμε πολύ σημαντικά στο Κοινοβούλιο για τα παιδιά που δεν είναι ακόμη καν έφηβοι θα πρέπει να ζήσουν ε, με ε, συνέπειε αυτή τη απόφαση απόφασης πολύ πιο μακροπρόθεσμα από ότι οποιοδήποτε από εμά. και πολλέ ενώσει δικαιωμάτων των παιδιών έχουν προσπαθήσει τώρα να προσπαθήσουν να υπάρξει αντιστάθμιση, διάλογο ε, με του ανθρώπου οι οποίοι συμμετέχουν στι διαπραγματεύσει. Πώ μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι που να αντέξει στο χρόνο. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα επηρεαστούν, οι νεότεροι από τις αποφάσεις αυτές, πώς μπορούν να έχουν οποιαδήποτε επιρροή ή άποψη για το τι θα γίνει. Και δεν το λέω αυτό μόνο λόγω των πανεπιστημίων και το που βρίσκονται το λέω και για το Erasmus Plus. Είναι επικίνδυνο, δεν αφορά μόνο το πανεπιστήμιο, μιλά, αφορά για τους απλούς ανθρώπους ε, οι οποίοι μέσω επίσημων και ανεπίσημων ε, ε, διαδικασιών συναντούν ένα τον άλλον. Κριστίνα Τιμπάτσκα και μετά θα κλείσω τις ερωτήσεις για αυτόν τον πρώτο γύρο γιατί θα έχουμε και άλλες δυνατότητε να συζητήσουμε. Κριστίνα. Ε, Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στον καιρό του ίντερνετ δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί κανεί. ούτε στον κόσμο των επιστημών, ούτε στον κόσμο του πολιτισμού. Οπότε οδηγούμαστε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Θα υπάρχει η δηλαδή η Λευκορωσία στον ευρωπαϊκό ε, χώρο, αλλά δεν θα υπάρχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, στην αρχή, ίσως ως προτεραιότητα, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αν θέλουμε και αν μπορούμε να διατηρήσουμε το Εράσμος και αν μπορούμε να διατηρήσουμε το χώρο επιστημών και έρευνας για το επόμενο ε, πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα καθώς επίσης και ε, τη συνεργασία στον ε, τομέα της, ε, των δημιουργικών τεχνών. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Έχετε το λόγο, κύριε Κατζάνο, για να απαντήσετε. Grazie. Σας ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις σας είναι όλες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα ήθελα να απαντήσω με ταχύτητα. Πρώτη ερώτηση. Το να έχουμε λοιπόν ένα κατάλογο με όλα. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη διαπραγμάτευση θα πρέπει ήδη να έχουμε εξαντλητικό κατάλογο γιατί δεν μπορεί να πούμε «Α, ξέρεις, ξέχασα το ένα ή το άλλο ή το τρίτο στοιχείο». Έχετε πολύ το δίκιο, πρέπει να γίνει ένας κατάλογος. Από την άλλη πλευρά από την άλλη πλευρά θα πρέπει, και αυτό είναι απόλυτη ανάγκη, ε, πρέπει να είναι διαφανής ο κατάλογος αυτός. Δηλαδή η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ε, ε, θα πρέπει να, να, να αποτελέσει η διαπραγμάτευση αυτή μια απλή διακυβερνητική ε, ε, σχέση και μια διακυβερνητική διαπραγμάτευση, πράγμα που ίσχυε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πριν αρχίσει να υπερισχύει το διεθνές δίκαιο. Θέλω να πω με αυτό ότι ο απλός άνθρωπος του δρόμου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο απλός πολίτης που όμως είναι Ευρωπαίος πολίτης, είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος με αυτήν την ιστορία του Brexit που είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Επομένως η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική, ο, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ σημαντική και επίσης πολύ σημαντική επίσης είναι η εργασία αυτών που προωθούν τα και θα προωθήσουν, θα κληθούν να ε, προωθήσουν τα αποτελέσματα. Γιατί από μία διαπραγμάτευση μπορεί να γεννηθεί, να προκύψει και κάτι θετικό. Διότι μπορεί να είναι αντιτιθέμενες οι απόψεις, ναι, αλλά είναι σημαντικό αυτές οι αντιτιθέμενες έστω απόψεις να είναι γνωστές σε όλους. Το κοινό να τις γνωρίζει τις απόψεις αυτές. Εγώ πραγματικά θα απογοητευτώ αν η διαπραγμάτευση γίνει κλειστή και σε καθαρά διακυβερνητικό ε, ε, επίπεδο. Ε, και είναι προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης θα πρέπει να κοινοποιήσει τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Λέω στην κυρία Σίλβια Κώστα ότι τα μέσα ενημέρωσης βεβαίως είναι ε, πολύ σημαντικό, από το ακουστικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό και από πλευράς οικονομικής επίσης, γιατί ε, ξέρετε η κουλτούρα, ο πολιτισμός δεν αφορά μονάχα κάποιους λίγους προνομιούχους ε, και όταν εγώ μιλάω με ερευνητές και όταν αναφέρομαι σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους μοναχούς, ε, τους πολύ οι έγκριοι τους, ε, του, του Μεσαίωνα που παίρναν το δισάκι τους και πηγαίναν από μοναστήρι σε μοναστήρι. Όχι, εδώ μιλάμε ε, για ε, την έρευνα. Εδώ λέμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε η, ας πούμε τα πολύ ακριβά ερευνητικά επιστημονικά περιοδικά να γίνουν ε, προσβάσιμα σε όλους. Όταν είναι επιγραμμικά διαθέσιμα γίνονται ε, πολύ πιο προσιτά. Και υπάρχει βεβαίως και το οικονομικό στοιχείο του copyright. Δεν είναι δυνατόν ε, να κλέψει κανείς το copyright και να διοχετεύσει και να προωθήσει διάφορα έργα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ψηφιακή αγορά, η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αφορά και τον γεωαποκλεισμό, που είναι η πρώτη μορφή ε, μέσα από την οποία μπορεί κανείς ε, να ακολουθήσει και σε άλλη χώρα τα στοιχεία ή τα, τις συμβολές τις έχει σε μία χώρα, να τις ακολουθήσει, εν και σε μία άλλη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα αναφέρω εδώ και την περιαγωγή, γιατί τώρα ξέρουμε ότι από 15 Ιουνίου και μετά, χωρίς καταχρήσει και με εύλογη χρήση, φυσικά ε, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ίδιο πρόγραμμα που έχει στη χώρα του και σε άλλες χώρες. Επομένω, τώρα τώρα ε, όντως ακόμα και για τις collecting societies ε, γνωρίζετε ποιες είναι ε, τα, είναι οι εταιρείες οι οποίες συλλέγουν ε, τα χρήματα από τα πνευματικά δικαιώματα μέσα από αυτές τις διαδικασίες όλες λέω και μέσα από τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προεκύψει από την ομολογία του δικαστηρίου και από τα νέα νομοθετήματα με όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης αποκτούν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αλλά μην ξεχνάμε ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε μια κοινή στέγη και θέλω να πω στη Σίλβια Κώστα ότι ενδεχομένως χωρίς και να μειώσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βεβαίως αποτελεί την καρδιά της Ευρώπης ε, να λάβουμε υπόψη μας ίσως και το Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, υπάρχει ε, μια σύμβαση η οποία είναι σχεδόν παράλληλη με την οδηγία για την τηλεόραση χωρίς ε, σύνορα ε, και κάνουν δουλειά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα. Η εξέλιξη των τεχνικών, η εξέλιξη ε, της τεχνογνωσίας και των επιστήμης και της επιστήμης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά ταυτοχρόνως να προστατεύονται και οι μικροί και οι ανήλικοι γιατί υπάρχουν ε, περιεχόμενα τα οποία παραβιάζουν ε, τους, ε, τις αρχές που διέπουν τους ανηλίκους. Δεν μου το ρωτήσατε, αλλά εγώ το, τονίζω. θα πρέπει οπωσδήποτε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό που είναι το ε, δραστηριότητες οι οποίες υποδαβλίζουν το ρατσιστικό ε, μίσος θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Η ελευθερία είναι, είναι ακριβώς ε, εκεί που οι ελευθερίες του ενός μπορεί να σκοντάψουν πάνω σε ελευθερίες άλλων. Ε, δεν λέω ότι θα πρέπει να καταργηθεί ε, η, ελευθερία της ε, κατάρτισης ή της εκπαίδευσης ή της έκφρασης, αλλά θα πρέπει να βρεθεί αυτή η χρυσή γραμμή η οποία είναι απαραίτητη και είμαι βέβαιος ότι μια και μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει μακρά και ισχυρή παράδοση στους τομείς που μόλις ανέφερα, θα βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο της συζήτησης. Ίσως ε, στο τέλος ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης να υπάρξει κάτι και να θέλετε και πάλι να παρέμβετε. Πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Να καλωσορίσω τον δόκτορα Τόμας Έκμαν Γιώργενσεν. Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων και θα μας δώσει μια γενική εικόνα για το ποιες είναι συγκεκριμένες επιπτώσεις του Brexit στα πανεπιστήμια. Τι συζητείτε, τι επιπτώσεις αναμένονται ε, και σε, και σε σχέση με, τον, ε, το πολύ αγαπημένο μας πρόγραμμα, το Erasmus. Δόκτωρ ε, Γιώργινσεν, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ε, για όσους δεν μας γνωρίζετε, είμαστε η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 850 ε, πανεπιστήμια, 30, 47 ε, χώρες. Βλέπετε εδώ έναν χάρτη που δεν σας δείχνει πόσοι είμαστε, πόσο μεγάλοι είμαστε, αλλά βλέπετε ο κόσμος της ανώτερης εκπαίδευσης πηγαίνει πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς είναι και πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει ολοκλήρωση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ πιο δύσκολο από την έρευνα, για παράδειγμα. Για να σας πω ποια είναι η δική μας άποψη για το Brexit, κατά τη γνώμη μας, το πάμε από την αρχή, η οικογένεια των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων πρέπει να παραμείνει ενωμένη το, τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη βεβαίως έχουν μια ιστορία που είναι μεγαλύτερη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά φυσικά δεν χαιρόμαστε να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει τη συνεργασία στο πανεπιστημιακό τομέα και βλέπετε ότι σύντομα αμέσως μετά το δημοψήφισμα ε, είχαμε μία διάσκεψη, ε, είχαμε 24, ε, διασκέψεις Πριτάνεων, οι οποίοι προσυπέγραψαν μία δήλωση ότι θέλουν να συνεργαστούν. Έχουμε ενημερωτικά δελτία για το τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Ε, εν ολίγης πιστεύουμε ότι μία εύκολη επικερδής για όλους ε, λύση είναι ε, η καλύτερη ε, συμφωνία σύνδεσης με τα, για τα επόμενα μελλοντικά προγράμματα Εράσμους και στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 χρειάζεται λίγη πολιτική θέληση αλλά αυτό χρειάζεται μόνο. Τώρα, το άμεσο ζήτημα, το άμεσο ζήτημα, όπως έχει υποθεί και στο παρελθόν, το άμεσο ζήτημα είναι η κινητικότητα των φοιτητών γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, κατά πολύ ε, ο, ο ε, ε, αγαπημένος προορισμός των Ευρωπαίων φοιτητών πάνω από 200.000 φοιτητές ε, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή θα ε, φοιτήσουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο άμα λάβει κανείς την υπόψη την κινητικότητα των πιστοποιητικών και των μονάδων. Νομίζω 120.000 είναι για τα πτυχία είναι πολύ λίγο, λίγο αυτό που μπορούμε να κάνουμε και να πούμε ότι α, ε, μπορούμε να ε, τα ε, φτιάξουμε τα πράγματα με καλύτερο τρόπο. Σχόλιο εκτός μικροφώνου δυστυχώς δεν το ακούσαμε. Ε, πάντως η απάντηση είναι ότι ναι, μπορείτε να χτίσετε βέβαια πολύ πιο ε, γρήγορα. Ε, το θέμα είναι πού θα πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα πρέπει να χτίσουμε νέους, ε, νέες φοιτητικέ. φοιτητικές. Λοιπόν, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Αν δούμε, ας πούμε, ότι θα είναι πολύ έντονο, θα είναι πολύ έντονη η ώρα της διαπραγμάτευσης και έτσι το Brexit ε, θα γίνει με τους χειρότερους όρους, υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, οι φοιτητέ να πρέπει να περάσουν πολύ δύσκολες και δαπανηρές διαδικασίες για να φοιτήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει επίσης η διαφορά μεταξύ των εγχώριων και διεθνών διδάκτρων, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε ότι ότι τα πράγματα θα είναι πιο σαφή στην επόμενη συνεδρίαση, στην επόμενη συνάντηση. Ε, θα γνωρίζετε ενδεχομένως την οδηγία 2016 801. Ε, ε, η Δανία δεν συμμετέχει, αλλά το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στην οδηγία. Η, αν έχει κανείς μία ε, σύμβαση, ε, αν μπορεί να πάει κανείς σε ένα πανεπιστήμιο, Μπορεί να φέρει την οικογένειά σου, να μείνει να εργαστεί υπό πολύ καλές συνθήκες. Ε, υπάρχει ε, νομίζω μία πολύ άνηση μεταχείριση και αυτό δεν είναι καλό για, καθέ, κανέναν. Ε, υπάρχει μία, διά, μία αυξανόμενη τάση χρήσης αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Έχουμε αυτό λοιπόν, το, αυτήν την πραγματική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 πρόκληση. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα ήθελε να, είναι, να, μπορούν να έχουν κινητικότητα, δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί δεν μπορούν να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως ενδεχομένως ε, οι Ιρλανδοί ε, να ε, τα ε, καταφέρουν κάποια στιγμή, αλλά βραχυπρόθεσμα θα υπάρξουν κάποιοι φοιτητέ που δεν θα μπορούν να ασκήσουν την κινητικότητά τους. Νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφάνεια για το Εράσμος η ε, Κριστίνη θα τα πει με περισσότερες λεπτομέρειες. Κανονικά, από νομικής απόψεως, είναι απλά τα πράγματα. Ε, μπορεί να είναι ε, μια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, που συμμετέχει στο πρόγραμμα. είναι πολύ σαφής η μέθοδος, απλή. δεν συνδέεται άμεσα με το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ε, όμως είναι πιο φιλικό για τον τρόπο με τον οποίο εμείς τουλάχιστον ως Ένωση λέμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε. Να υπάρχουν εθνικοί φορείς ε, για το ε, Εράσμους. Υπάρχουν ε, κάποια σημεία ενημέρωσης στην Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με αυτό. Οι Βρετανοί όμως δεν θα θεωρήσουν ότι θα μπορούσε να γίνει ε, εύκολα η επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο έδαφο τους. Δεν θα το πάρουν πολύ καλά αυτό, γιατί ακριβώ υπάρχουν αυτοί οι εθνικοί φορείς και φαίνεται ε, πολύ πιο ε, δύσκολα αυτά που πρέπει να υπογράψει κανείς για το Εράσμου σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο πώ ήταν τα πράγματα πιο πριν και όχι να γίνονται όλα μέσω των εθνικών φορέων τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφάνεια. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα. αν ακολουθήσει κανείς κατευθυντήριες γραμμές ε, της, ε, της διαπραγματευτικής ομάδας, τότε είναι πολύ μεγάλος, πολύ ψηλά ο πύχης ε, για κάποιον ε, που γεννιέται από Ευρωπαίους γονείς ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2009 το Μάρτιο θα έχει πρόσβαση στο Βρετανικό επαιδευτικό σύστημα σαν να ήταν Βρετανός πολίτης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το θέμα των διδάκτρων θα ήταν πάρα πολύ επωφελές, πιστεύουμε ότι είναι καλό βέβαια, γιατί θέλουμε ευρωπαϊκή πρόσβαση στο ε, βρετανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υπάρχει λόγος για τον οποίο όλος ο κόσμος θέλει να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι μόνο το θέμα των Αγγλικών, αλλά και γιατί το βρετανικό εκπαιδευτικό ε, περιβάλλον είναι πάρα πολύ καλό και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό και ελπίζαμε λοιπόν να υπάρχει ένας πολιτικός τρόπος από πλευράς Βρετανίας και από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί ένας συμβιβασμός γιατί δεν θα υπάρχει ένα πρόβλημα διακριτικής μεταχείρισης, κατά πόσο γίνεται διάκριση εναντίον των ε, ε, Ινδών, για παράδειγμα, και υπέρ των Ισπανών. Ε, Νομικό, σε πάση περιπτώσει, είναι ένα δύσκολο, περίπλοκο πρόβλημα. Επίσης έχουμε την αναγνώριση, την αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στις ε, διαπραγματευτικές κατευθυντήριες γραμμές σαφώς. Δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που παίρνουν την αναγνώριση. Ε, δεν γίνεται αναγνώριση ενός γιατρού, ας πούμε, του δίνουμε μια δουλειά στο νοσοκομείο και τον Απρίλιο του 2019 του λέμε «Α, δεν ισχύει αναγνώριση πια, αυτό δεν νομίζω να συμβεί» θεωρητικά είναι πιθανό, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Λογικά πρέπει να υπάρχει επαγγελματική αναγνώριση. Μιλάω μόνο για την επαγγελματική αναγνώριση, η οποία διέπεται από την οδογία. Τώρα η ακαδημαϊκή αναγνώριση, ε, επόμενη διαφάνειά μου, είναι ε, η ε, αποσύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του EHEA, Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο αποφάσεων που έχει να κάνει με, τον κανονισμό, με τους κανονισμούς που αφορούν το Εράσμους. υπάρχει επίσης ε, ένα θέμα ε, διαπραγμάτευσης που αφορά το ε, ET 2020 και η διαδικασία της Μπολόνιας, δηλαδή διακυβερνητικές διαδικασίες που ισχύουν επίσης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αν δει κανεί, για παράδειγμα, το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων, αν δει κανεί το ECTS. Ε, θα ήταν λοιπόν προτιμητέο για όλους, ε, πιστεύουμε, να, είναι, να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και από τη Βρετανική και από την Ευρωπαϊκή πλευρά για να συμμετέχουμε στην μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού, στη διακυβερνητική μέθοδο, για να υπάρξει ένας διακανονισμός υπέρ ενό σεναρίου που όπως είπα από την αρχή θέλουμε να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη Μεγάλη Βρετανία. Πάντω είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Η νομοθεσία είναι δύσκολη, αλλά όχι τόσο περίπλοκη ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί από το θέμα των πανεπιστημίων με λίγη καλή πολιτική θέληση. Ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δόκτωρα Γιώργενσεν. Βεβαίω θέλουμε να ακούσουμε και τη βρετανική ε, άποψη, γιατί αυτοί είναι που θα πληγούν κυρίω από τι ε, συνέπειε, οπότε να ε, καλωσορίσω την καθηγήτρια Κριστίνα Σλέιτ. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η αναπληρώτρια πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μπαθ. Very much, Chair, and thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ε, πρόσκληση. Και ευχαριστώ, Τόμας, που ήσουν τόσο θετικό για το Εράσμους, γιατί και εγώ ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω. Όλα τα πολιτικά χρήματα είναι ιδιαίτερω παγκοσμιοποιημένα, αλλά τα, τα πανεπιστήμια πάντα ήταν παγκοσμιοποιημένα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό, να μην περιορίζεται η γνώση από σύνορα. Για μένα, και αν ε, ακούσετε θα καταλάβετε ότι είμαι και Αυστραλή εκτός από Βρετανίδα. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης ήταν το Εράσμους. Ο τρόπος που δημιούργησε αυτές τις, ε, αυτούς τους συνδέσμους που κατέστησαν τη ζωή των φοιτών πολύ καλύτερη. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι φοιτητέ χρειάζονται πολύ περισσότερο, περισσότερο από ποτέ τα δίκτυα που προκύπτουν από τις σπουδές στο εξωτερικό. Και θα συνεχίσω να μιλώ για το θέμα αυτό έχει να κάνει και με τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες. Σε αυτούς τους ε, τομείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι ώστε να έχουμε ε, άτομα που μπορούν να βρίσκονται στο Μέχελεν και να συνεργάζονται με κάποιον στην Κίνα. Αυτό πρέπει να το προωθήσουμε και για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Θα μιλήσω για το Erasmus Plus, αλλά θα επικεντρωθώ σε κάποια κομμάτια μόνο, στην κινητικότητα και σε αυτό που κάποτε ονομαζόταν τέμπους και η δυνατότητα, η δημιουργία μάλλον δυνατοτήτων, ε, η δράση κλειδί 2. Ως ε, αντιπρίτανης και ως Βρετανίδα βεβαίως και εγώ, αλλά και εσείς πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Μια, ένα από τα λυπηρά για την Βρετανία είναι το επίπεδο της κινητικότητας των ε, φοιτητών. 7% το 2014-2015. Η Βρετανική κυβέρνηση βεβαίως θέλει να αυξήσει το ποσοστό αυτό, αλλά σκεφτείτε πόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό αυτό από άλλες χώρες. 15% στις ΗΠΑ, 19% στην Αυστραλία, 25% των Γερμανών φοιτητών είναι σε προγράμματα κινητικότητας ως προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Και εγώ δουλεύω ε, με, την, ε, με το Πανεπιστήμιο στο Μεξικό και λένε ότι έχουν 80% ε, στο, είχαν 80% κινητικότητα από τους φοιτητές, έχουν στόχο τώρα να το φτάσουν αυτό στο 100%. Και το ίδιο ισχύει για τα κινέζικα πανεπιστήμια. Οπότε δεν είναι ότι είμαστε και στι πρώτε θέσει. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Και στην Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε. Το... Είναι καλό το αφήγημα αυτό για το ότι το Εράσμος είναι... έχει αποδειχθεί επιτυχές, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτά τα στοιχεία εδώ είναι γνωστά και βλέπουμε ότι Λιγό, λίγοι φοιτητέ ε, είναι σε προγράμματα ε, κινητικότητα, αλλά όποιοι είναι έρχονται κυρίω στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η βρετανική άποψη. Το άλλο που είπατε, είπες και εσύ, είναι τα μεγάλα, οι μεγάλοι όγκοι ε, Ευρωπαίων φοιτητών που πάνε στην, στην στο Ηνωμένο Βασίλειο. 30.183 φοιτητές στα πλαίσια του Erasmus Plus. Χωρί να μιλάω για του άλλου 60.000 φοιτητέ οι οποίοι έχουν, ε, βρίσκονται σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι τεράστια λοιπόν η, ο αριθμό των φοιτητών που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτέ οι συνδέσει σε όλη την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Αυξάνουν τι ε, συνέργειε. οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν καλύτερα αγγλικά, γίνονται κομμάτι του αγγλόφωνου κόσμου. Εμείς επίσης στη Βρετανία μπορούμε να μάθουμε πολλά από τους Ευρωπαίους. Και ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της ε, διαδικασίας με τον Brexit είναι ότι οι περισσότεροι όταν ψήφισαν κατά του Brexit δεν ψήφισαν κατά του να έχουν την ταυτότητα του Ευρωπαίου στην ε, όλη κουλτούρα των δυτικών ε, πανεπιστημίων ή τουλάχιστον ελπίζω η ευρωπαϊκή λοιπόν ε, ταυτότητα που δημιουργούμε και που προωθούμε μέσω αυτών ακριβώς των συνεργασιών και βεβαίως υπάρχουν ε, ε, πολλά που μπορούμε να πούμε είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η έρευνα που γίνεται στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Τώρα για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Το πανεπιστήμιο από το οποίο έρχομαι εγώ δεν εκπροσωπείται πολύ συχνά. Είναι μικρό α, πανεπιστήμιο. Αλλά βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο που ανήκει στην, στο Δουκάτο του Κόρν, στην Ουαλία. Και έχουμε αυτή την, αυτή τους ε, φοιτητές που ε, βρίσκονται στην, σε ένα πρόγραμμα διευρυμένης συμμετοχής, ε, χαμηλών εισοδημάτων, με λίγες ευκαιρίε. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνειδητοποίησα λίγο αργά ότι το είδος της κινητικότητας που εσείς εδώ, η δική μου οικογένεια, οι οικογένειες των παρισταμένων εδώ θεωρούν ότι είναι φυσιολογική, δηλαδή η πιο κοινή ερώτηση που έκανες Εράσμος, που σπούδασε στο εξωτερικό, που έκανε το εξάμεινο των ε, ε, σπουδών στο εξωτερικό, είναι, πολύ, είναι τελείως ξένο για πολλούς, γιατί πολλοί δεν έχουν αυτή την, ε, πολιτιστική πρωτεύουσα που τους κάνει να αισθάνονται άνετα ακόμα και δεν είναι στη χώρα τους. Πολλοί από τους δικούς μας συζητητές φοβούνται να πάνε στο Λονδίνο. Εντάξει, βέβαια αυτό ίσως και να είναι λογικό. Αλλά εδώ βλέπετε τι μας είπε μια, φοιτητριά μας που ε, ε, σπούδασε στο εξωτερικό. Είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να φύγει από το σπίτι της, ήταν αφοβισμένη, αλλά έκανε τελικά τεράστια διαφορά στη ζωή της. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της. Και αυτό που ξέρουμε και ε, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ ανθεκτικά αποτελέσματα που μας δείχνουν ότι για αυτούς που έρχονται από, οικονομικά, από περιορισμένα οικονομικά περιβάλλοντα και ευκαιρίες είναι πολύ σημαντικότερο να σπουδάσουν στο εξωτερικό από αυτούς που έχουν καλύτερο υπόβαθρο. next point I to, to mention just briefly. Oh, this, so here's the... Πάμε τώρα στα, στην διαφάνεια για τα ωφέλη της κινητικότητας. Προφανώς είναι σαφή όλα, αλλά αυτό που έχουμε εμείς ως ε, θεματολόγιο και ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ είναι ότι θέλω να σας πω ότι όλοι Ευρωπαίοι, Βρετανοί, όλοι πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην χάσουμε κάτι τόσο πολύτιμο. Μπορεί να είναι δύσκολο, περίπλοκο, Μπορεί να, πώς το είπε ο Τόμας, να, να χτενίσουμε λίγο κάποια σημεία της νομοθεσίας. Ό,τι και αν είναι πρέπει να το κάνουμε. Εδώ βλέπετε εμένα στο Κίεβο για τη δημιουργία δυνατοτήτων. Πήραμε μια ομάδα στο α, Κίεβο, στο ε, Πανεπιστήμιο Τάρας Ναυτσένκο και ήταν πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο που ε, είχε εξειδίκευση στην ε, κατασκευή των ε, μηχανικών συστημάτων για τους δορυφόρους για την, που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι. Κάνουμε λοιπόν πολλή δουλειά με το Πανεπιστήμιο του Κιέβου και νομίζω ότι αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές διαδικασίες και πρέπει να τις συνεχίσουμε. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε δεν θα πω πολλά ακόμη, αλλά θα πω ότι ως ε, επικεφαλής ενός πανεπιστημίου θέλω να πω ότι ε, ε, εξ όλων των πανεπιστημίων πόσο πολύ εκτιμούμε το Erasmus, το Erasmus Συν, το πόσο πολύ περήφανοι είμαστε ότι μπορούμε να είμαστε κομμάτι μια, ενός πολύ σημαντικού εμπορικού ονόματος και πρέπει να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε αυτά τα περίπλοκα θέματα. Γιατί ναι, οι πολίτες είναι και, μετακινούνται και εκτός Ευρώπης και υπάρχουν μοντέλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε και πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Ας διατηρήσουμε λοιπόν αυτές τις ε, σχέσεις που έχουμε. Ας μην, τις, ας τις αφήσουμε να ε, εξαφανιστούν. Θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, ε, ένθερμη παρέμβασή σας. Είναι σαφές ότι και για τα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι πολύ ε, σημαντική η ανταλλαγή αυτή με άλλα πανεπιστήμια. Θέλουν να συνεχιστεί έτσι ώστε και οι Βρετανοί φοιτητές να μπορούν να υποφεληθούν από αυτή τη σημαντική εμπειρία να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε και πάλι από τον κύριο Στρογεύσκη. Ένα λεπτό και πάλι σας το υπενθυμίζω. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας διότι πραγματικά μιλήσατε λες και είσαστε μέλος της Επιτροπής μας. Θα μπορούσατε να είσαστε πρέσβυρά μας. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, ήθελα να αναφέρω μονάχα δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρώτον, να θυμίσουμε ότι εκτός από το Erasmus Plus υπάρχουν και νέοι οι οποίοι μελετούν χωρίς όμως να συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, αλλά είναι ένα, μια μεγάλη ομάδα η οποία μετακινείται ε, ιδιωτικός κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε. Ε, πρέπει να τους λάβουμε και αυτούς υπόψη. Ναι. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Στην Ευρώπη Υπάρχουν ιστιτούτα όπως το Θερβάντες, όπως το Γκέτε, όπως το British Council, το Βρετανικό Συμβούλιο. Ποια θα είναι η μοίρα του British Council μετά από το Brexit και κάτι τρίτο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε άλλες συμφωνίες και σε άλλες νομοθετικές πράξεις ε, έχει γίνει λόγος και ε, για ε, διπλή φορολόγηση των εργαζόμενων στον τομέα του πολιτισμού. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να διευθετηθούν τα ζητήματα αυτά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα με διπλές πληρωμές και διπλούς φόρους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέλλη. Έχετε το λόγο κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τους δύο καλεσμένους μας. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, όπως και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Υπάρχουν αυτοί που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί που θέλουν πραγματικά να μείνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικοί μάλιστα περισσότερο και από άλλους. Υπάρχει ένα σενάριο ε, που μπορεί ίσως να θεωρηθεί σαν κορφολόγημα, cherry picking, διαλέγω τα καλύτερα, αυτά που μου αρέσουν. Ο κύριος Φερχόφστατ ε, το είχε αναφέρει αυτό, είπε ότι δεν θα, ε, δεν θα δοθεί η δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να κορφολογήσει τα καλύτερα. Εσείς πώς το βλέπετε εσείς λέτε ότι το Brexit είναι Brexit όταν λέμε φεύγουμε είναι φεύγουμε ή υπάρχει κάποια πορτούλα ανοιχτή για το cherry picking. Τι θα γίνει κυρίως εάν ε, η Βρετανική πλευρά ε, υιοθετήσει το hard Brexit. Ευχαριστώ πολύ. for your commitment to... Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας ε, και γιατί ξεκαθαρίσατε για μία ακόμα φορά πόσο, σημαντικές, πόσο σημαντικά συγγνώμη, είναι τα προγράμματα ανταλλαγών για τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές όλα τελικά εξαρτώνται, εξαρτώνται συγγνώμη, από την πολιτική βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή κατά πόσον ε, θα αποφασίσει να συνεχίσει τουλάχιστον να πληρώνει για τα χρήματα αυτά στον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. Δεν τα ξέρουμε ακόμα. Η, τι θα γίνει όμως ε, με τους ε, φοιτητές σας, ε, θα προσπαθήσουν και αυτοί να ακουστεί η φωνή τους, να πούνε ότι τους ενδιαφέρουν τα προγράμματα αυτά, ότι τους ενδιαφέρει να μην σταματήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις οι οποίες εστίασαν ακριβώς στα ζητήματα τα οποία ε, αντιμετωπίζουμε που έχουμε μπροστά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς γιατί μιλήσατε αγαπητή κυρία με μεγάλο πάθος. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο την περίοδο μέχρι το 2019 οπότε πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί εμείς ε, ζητήσαμε σαν προϋπόθεση από πλευράς της Ευρώπης και από πλευράς της Ευρωπαϊκής του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνουν ε, εξ αρχής σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης που ζουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και των ε, πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρώπη. Μιλάμε μετά το 19 τώρα κυρίως τι θα γίνει. Ο Καθηγητή ε, Κατζάνο μίλησε προηγουμένως για διαφάνεια και η κυρία Τρούπερ, συνάδελφός μου, αναφέρθηκε στη θέση των ε, ε, ίδιων των φοιτητών. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι οι σχέσεις, ενδεχομένω, ποιε είναι οι κινήσεις του εκπαιδευτικού, ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών, με την κυβέρνηση, με τους βουλευτές, έτσι ώστε να ε, προωθηθεί ας πούμε αυτό το περιβόητο νορβηγικό μοντέλο. Τελευταία ερώτηση. Σε πολλές ε, περιπτώσεις, ε, μάλλον συγγνώμη, ο τρόπος με τον οποίο ψήφισαν οι νέοι είναι σαφές μετά από ανάλυση ότι ήθελαν τον Remain και όχι τον Brexit. Άρα στι συζητήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο ή ε, το, το, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σεβαστεί αυτούς τους νέους. Γιατί δεν έχουμε μόνο το Εράσμους, έχουμε και το, ε, ε τις θελοντικές ε, διαδικασίες, έχουμε ένα σωρό προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφο Σοντρόβα. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο το, της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στη δική σας, στο επίπεδο της δικής σας ε, οργάνωση, γιατί εκπροσωπείτε πάνω από 850 πανεπιστήμια, ίσως, ε, ίσως λέω, θα μπορούσατε ας πούμε να κάνετε μια κοινή δήλωση statement ή declaration για το τι θα θέλατε μετά από το Brexit ή το πώς θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα έρασμος μετά το Brexit ή κάτι τέτοιο. Γιατί κατά την άποψή μου και τα πανεπιστήμια μπορούν να κάνουν, να ασκήσουν πίεση, είναι, μπορούν να είναι καλά σε, στο, σε διαδικασίες lobbying. Άλλωστε, η αντιπριτανη ε, ε, αναφέρθηκε κάπως στο θέμα αυτό. Ε, πάντα τα πανεπιστήμια λένε ότι είναι πολύ σημαντικέ και οι μεμονωμένε σχέσει με, ε, με άλλα πανεπιστήμια. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και στο μέλλον. Μιλάω για τους φοιτητές που βρίσκονται στο βάθος της αίθουσας που τους κάλεσα εγώ ε, και ανα, ξέρουν κάτι που το ξέρω και εγώ. Εγώ ήμουν καλλιτέχνης πριν από ε, την πολιτική μου καριέρα και ξέρω, δουλεύοντας με πολύ κόσμο από όλη την Ευρώπη, πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους καλλιτέχνες. Ανησυχούν πάρα πολύ για τις ε, δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Το ερώτημα λοιπόν των φοιτητών είναι έμαθαν τη σημασία των ε, δημιουργικού, του δημιουργικού κλάδου και πόσο βοηθά, πάρα πολύ, πόσο βοηθά η κινητικότητα και η προσβασιμότητα. Όμως, ε, πόσο το επιχειρηματικό πνεύμα της ε, νεολαίας θα επηρεαστεί από το Brexit και τι κάνουν τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου για να διατηρηθεί αυτό το πνεύμα. Ευχαριστώ. Το τελευταίο ερώτημα είναι ερώτημα μάλλον θα μπορούσαν να, να απαντήσουν οι, οι στο τελευταίο πάνελ που είναι εδώ ακριβώς για τον ε, τομέα του πολιτισμού και των ε, δημιουργικών ε, βιομηχανιών. Να δώσω το λόγο και στους δύο εμπειρογνώμονες, την, καθη... την καθηγητή Σλέιτ και τον κύριο Γιώργενσεν. Αν μπορείτε όσο πιο σύντομα γίνεται, έτσι ώστε να έχει και το τρίτο πάνελ επαρκή χρόνο. Έχετε το λόγο, όποιος θέλει μπορεί να ξεκινήσει από τους δυο σας. I'm going to propose to say a little about the young, young... Θα ήθελα και εγώ να πω μερικά πράγματα για τους νέους. Δεν έχω απάντηση για τη διπλή φορολόγηση βέβαια. Ε, θα το αφήσω εσένα, ε, για εσένα την, το διαλέγουμε και παίρνουμε, ε, Τόμας, εσένα θα το αφήσω. Ε, νομίζω ότι και εσύ είσαι σε θέση να μιλήσεις για την πολιτική βούληση. Ε, ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ερώτηση των φοιτητών ε, και αν αρχίσουμε με την ιδιωτική κινητικότητα. Η ιδιωτική κινητικότητα του Ινστιτούτου Γκέτε έχει δουλέψει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και έχουμε και εμείς ε, φοιτήσει σε άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δούλευε μια χαρά. Ε, δούλευε και χωρίς το Εράσμους και αυτό μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει και δεν βλέπω να υπάρχει κανένας λόγος ούτε πιθανότητα να σταματήσει αυτό τα μεγάλα ζητήματα, σπουδαία ζητήματα, αυτά τα οποία δεν ετέθησαν είναι πώς τις μεταφορές των ε, μονάδων από τα μαθήματα μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι παρόλα αυτά όμως και παράλληλα συναρπαστικό. Ποιες είναι οι προοπτικές Τη δημιουργία ενός κόρου που θα μπορούσε να είναι τόσο ζωτικό και ε, τόσο ε, δυναμικός, ίσως κάποιοι να θυμούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικό, σημαντική συμβουλή του στην δημιουργική κινητικότητα. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί με την κινητικότητα που είχαμε και είναι στο χέρι μα να εξασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό. Ε, όσον αφορά αφορά το να ψηφίζουν οι νέοι. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάνε να ψηφίσουν οι νέοι. Αυτή η διαδικασία που εξελίσσεται ε, μας οδηγεί στο να πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι το ότι γυρίζουμε πίσω σε παλιές ε, ερωτήσεις, αλλά να μην χάσουμε όλα αυτά ε, τα αξιέπαινα πράγματα που έχουμε επιτύχει ως τώρα. Έχεις εσύ το λόγο, Τόμας. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν θα μιλήσω για το διαλέγω και παίρνω, το cherry picking. Ε, δεν είναι ένα τομέα στον οποίο ενθαρρύνεται το να διαλέγουμε και να παίρνουμε. Ε, υπάρχει στους κανονισμούς, υπάρχουν διατάξεις στους κανονισμούς για την συμμετοχή τρίτων χωρών ε, πάρα πολύ σαφές διατάξεις. Ε, το να διαλέγει και να παίρνει κανείς δεν είναι πάρα πολύ καλό όταν είναι κανείς ε, έξω, όσο, όταν είναι μέσα. Ε, έχεις να παρουσιάσεις ένα, έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόγραμμα και ένα λογαριασμό και ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν με το αν είσαι έξω, αν και αν είσαι μέσα. Ε, αν θέλει λοιπόν κανείς να διαλέξει και να πάρει, ε, νομίζω ότι ε, στο λόγο, ε, στο Λάνκαστερ ήταν σαφές αυτό, θα ήταν περίεργο, υπόθηκε, ειδικότερα στους κανονισμούς που προβλέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών να μην υπάρχει μια ρήτρα για τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα για το ερώτημά σας που αφορά τους, την, την Ένωση Πανεπιστημία, πανεπιστημίων, ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, έχουμε κάνει ε, επανειλημμένως δηλώσεις μετά το δημοψήφισμα κάναμε ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέραμε συγκεκριμένα ε, για το Erasmus ε, Plus όπως επίσης και τον ορίζοντα 2020 που παραμένουν ανοιχτά για βρετανική συμμετοχή. Ε, όλα τα πανεπιστήμια γνωρίζουν ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εμείς βασιζόμαστε στην συνεργασία και στο ανοιχτό πνεύμα ε, αν θεωρείτε ότι χρειάζεται να γίνει μία ακόμη δήλωση, να κάνουμε κι άλλη μία. Όσον αφορά την ιδιωτική κινητικότητα, ναι, έχει λειτουργήσει, αλλά έχει λειτουργήσει γιατί υπήρχαν τα δικαιώματα των πολιτών και συνεπώς υπήρχε πρόσβαση στα δίδακτρα ε, σε ίδιο επίπεδο με τους Βρετανούς πολίτες. Το ερώτημα είναι αυτό θα λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν τα δικαιώματα αυτά και με την ε, αυξανόμενη παροχή μαθημάτων σε αγγλική γλώσσα σε άλλα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ελπίζουμε πάντως τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ε, τμήμα αυτής της, ε, ε, αυτού του, του ευρύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Πρέπει να περάσουμε άμεσα στο επόμενο πάνελ, αν θέλετε σύντομα, κύριε Κατζάνο. Ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι εάν δεν υπάρξει εσωτερική αγορά, θα υπάρξει ένα πρόβλημα εγκατάστασης των Αγγλικών Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η London School of Economics, ας πούμε, έχει έδρα στη Ρώμη, ας πούμε. Έχει παράρτημα. Ε, αυτό δεν θα είναι δυνατόν πλέον. Ε, θα πρέπει να γίνει ένα μοντέλο κεντρικού πανεπιστημίου. Ε, ε, ξέρετε ότι ε, υπάρχει πρόβλημα στην Ουγγαρία με το παράρτημα Αμερικανικού Πανεπιστημίου, επί του οποίου μάλιστα θέματος πήρε θέση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί και αυτό λοιπόν, μια τέτοια παρόμοια κατάσταση είναι σημαντική και πρέπει να την εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο σε έναν τομέα που είναι εξίσου σημαντικός, όπως και το Erasmus Plus, ο τομέας του, του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα, στον οποίο θα έχει επίσης ε, συνέπεια στο Brexit, οπότε ε, χαιρετίζω τον κύριο Μπέρντ Φέζελ, τον πρόεδρο του European Creative Business Network, το οποίο στα επόμενα 10 λεπτά, ο οποίος στα επόμενα 10 λεπτά θα μας παρουσιάσει το δίκτυό του καταρχάς και μετά θα μας μιλήσει για το τι κατά την άποψή του σημαίνει το Brexit για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού και της, ε, των δημιουργικών ε, βιομηχανιών. Έχετε το λόγο κύριε Φέζελ. Well, thank you, um, to the... Ευχαριστώ την Επιτροπή εγώ είμαι από το δίκτυο ε, των κλάδων των δημιουργικών και των πολιτιστικών. Βασιζόμαστε στο Ρότερνταμ, ε, έχουμε την έδρα μας στο ε, Ρότερνταμ, 41 μέλη όπως Εθνική φορείς, το Creative England, Creative Austria, τα οποία δημοσίως χρηματοδοτούνται από, από 19 χώρες, 70% του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δημιουργικού κλάδου εκπροσωπών πούμε 12 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, 75 ε, ε, συνολικής, ε, του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, 9 δις της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. αν, δείτε κανείς, λοιπόν, αν δει κανείς λοιπόν τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, νομίζω ότι ε, μπορούμε να πούμε ότι ο τομέας μας δεν έχει συμμετάσχει ούτε ε, έχει τύχει μεταχείρισης με διαφάνεια και ε, ισοτιμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως παίρνει η ο αντίστοιχο φορέας στην Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα. Θα ήθελα να αναφερθώ στον αντίκτυπο τώρα τι σημαίνει το να χάσουμε τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο τι σημαίνει να χάσουμε τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τι γίνεται με το εσωτερικό δυναμικό ε, των ε, ευρωπαϊκών, ε, του ευρωπαϊκού κλάδου αυτού προκειμένου να αντισταθμίσει το, την ζημιά ο ευρωπαϊκός δημιουργικός και πολιτιστικός τομέας δεν μπορεί να χάσει <clears throat> ούτε να αντισταθμίσει εύκολα την απώλεια. Ε, το ΑΕΠ είναι 95, ε, το, το ποσό 95 δις. Ε, πρόκειται λοιπόν για 20% ε, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε, λοιπόν, οποιαδήποτε, αντίκτυ, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αντίκτυπος υπάρχει είναι τεράστιος και σας το λέω αυτό και το λέω και σε σχέση με το διαλέγω και παίρνω. Είναι προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει, να διαλέξει αυτό ακριβώ το σημείο. Το δημιουργικό τομέα από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να το χάσει. Ενώ υπάρχουν λοιπόν και άλλα προγράμματα όπω το Εράσμου, όπου εξακολουθούν ε, μέχρι το 2019, το 2020. Εδώ, λόγω ε, της ε, συναλλαγματικής ε, ισοτιμίας και της απώλειας αξίας της λίρας χάνουμε από τις εξαγωγές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποια κράτη-μέλη αναμένουν 1% μείωση εσόδων το 2016. Κάτι αυτό, αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσει και κατά τα επόμενα έτη. Αυτή η μείωση εσόδων λοιπόν ισχύει ειδικότερα για μικρότερες επιχειρήσεις που δεν είναι παγκόσμιες αλλά εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορούν να αποσβέσουν με κάποιο τρόπο αυτό τον κίνδυνο 95% των χωρών της Ευρω... των ε, εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δημιουργικό ε, τομέα έχουν κάτω από 10 υπαλλήλους. Αυτός ο κίνδυνος λοιπόν που λαμβάνει τώρα χώρα αυτή τη στιγμή επηρεάζει τη μεγάλη πλειοψηφία των μικρών εταιριών στο δημιουργικό κλάδο. Είναι λοιπόν λογικό να λέμε ότι χρειαζόμαστε κάποιου είδους ε, ε σλόγγαν ε, κατά ε, ε, του κινδύνου από τον Brexit, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει να καταγράφουμε απώλειες. Επίσης, όσον αφορά την απώλεια εξαγωγών, οι περισσότερες εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8 δις ευρώ το 2012 που είναι η πιο πρόσφατη αριθμή και ο δεύτερος ε, εισαγωγέας ε, είναι με 5 δις ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες και ένα δις μόλις η Κίνα. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συμβεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει λιγότερα, το μισό ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη υπολόγισαν ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια κάτω χώρες, για παράδειγμα, πάνω από 16 δις ευρώ ετησίως, ε, αν η μείωση είναι περίπου 10% και αυτό είναι μόνο εκτίμηση βάσει των εμπορικών σχέσεων που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή και δεν ε, υπάρχουν στοιχεία και για την ε, έρευνα. Αλλά έχουμε πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης 6,1% των ε, θέσεων εργασίας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι Ευρωπαίοι ε, πολίτες, είναι πολίτες της Ένωσης 2% λοιπόν του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται αν δεν μπορεί να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κίνδυνος 240.000 θέσεων εργασίας που μπορεί να επηρεαστούν από αυτή τη σχέση των εργαζομένων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως αυτή η σχέση δεν είναι βαθμιαία, δεν είναι προοδευτική, ε, γιατί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι τομεί του δημιουργικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσαν να κάνουν αίτηση για θεώρηση. Δεν είναι μόνο θέμα κόστου, δηλαδή, είναι μια απαγορευτική διαδικασία. Η κινητικότητα λοιπόν ε, των ταλέντων είναι ε, πάρα πολύ σημαντική και, και της δημιουργικότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες εξαιρέσει ε, για τις θεωρήσεις, για τις εταιρείε κάτω των 10 εργαζομένων που είναι το 10% του τομέα μας. Τι θα γινόταν αν είχαμε λιγότερες εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 42% είναι όλων των ε, υπηρεσιών ε, που εξάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των δημιουργικών, του δημιουργικού κλάδου. Δεν υπάρχουν όμω μόνο εισαγωγέ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως προς αυτό το τομέα. Είναι και βιομηχανία, είναι ο τομέα τη υγείας όπω γνωρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα δημιουργικό κόμβο και το ερώτημα είναι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτό το καινοτόμο, την καινοτόμο συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο ζητήματα συνδέονται με αυτό το θέμα για να διατηρήσουμε αυτά τα ωφέλη από τις εισαγωγές. Πρώτον, είναι μια συνεκτική στρατηγική για την αντιστάθμιση της ενδεχόμενης απώλειας υπηρεσιών δημιουργικού κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ένας κλάδος που βασίζεται σε φορολογικές ελαφρύνσεις μέσω πολλών προγραμμάτων και πολύ διατομεακή διακυβέρνηση. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το Υπουργείο ε, Ψηφιοποίησης και Εκπαίδευσης. Λοιπόν, υπάρχει ανάγκη μιας διατομεακής προσέγγισης και για να υπάρξει αντιστάθμιση της ενδεχόμενης απώλειας, το Ευρωπαϊκό, ε, το Ενωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να μάθει από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον τομέα. Επίσης το θέμα της, ε, της, ψηφιακής ενιαίας, της αγοράς. Ο δημιουργικός κλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της ε, ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τις χώρες, για τις εταιρείες της τεχνολογίας. μία από τις κόκκινες γραμμές ε, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να συμμετέχει και να έχει άποψη για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό πρέπει να είναι από τις βασικές προτεραιότητες των διαπραγματευτικών ε, ε, διαδικασιών, να κρατήσουμε ανοιχτές τις αγορές και τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. Τέλος, μιλούμε πολύ συχνά για τα, τους δασμούς, ε, απώλεια, μάλλον απουσία ε, δασμών, όμως ε, ο δημιουργικός κλάδος που ανθεί εξαρτάται όχι μόνο από τους διαθρείς πυλώνες, αλλά και στην αστική διάταση, την αστική οικολογία, για να το πω έτσι, είναι λοιπόν και προς το μέγιστο όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μια αστική διάσταση που να ανθεί ε, στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ε, στι απαιτήσει του Ηνωμένου Βασιλείου για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα 8 δις που θα επενδυθούν στις πολιτιστικές δημιουργικές υποδομές των Ηνωμένων Βασίλειων, χαθούν αυτά τα χρήματα, θα είναι αρνητικός ο αντίκτυπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν ε, για τον αντίκτυπο του 20% ε, ε, που θα μπορούσε να, να σημάνει απώλεια. Ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να αυξήσουμε το εσωτερικό δυναμικό του δημιουργικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα το Δεκέμβριο του 2016 για του βασικού τομεί στου οποίου μπορεί να γίνουν επενδύσει. Θα σα πω μερικού, ε, θα διαλέξω λοιπόν και εγώ και θα πάρω πέντε που είναι σημαντικέ. Ένας, ε, η διαμόρφωση πολιτικής. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς διατομεακή εγκάρσια ευρωπαϊκή στρατηγική με την DG Growth, την DG Innovation και την DG Culture. Αυτό είναι κάτι το οποίο απουσιάζει αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται μια οριζόντια προτεραιότητα για του δημιουργικού κλάδου σε άλλα προγράμματα χρηματοδότηση τη Ένωση, σε παράδειγμα τον ορίζοντα 2020. Πρέπει να ανοίξει επίση και να αυξηθεί ο προπολογισμό του Creative Europe και της, ε, ε, του Guarantee ε, Facility. Όλα αυτά είναι βήματα τα οποία θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν, να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που διατρέχουμε. Τελευταίο θέμα Νομίζω το καλύτερο Brexit ε, θα ήταν καθόλου Brexit όσον αφορά τον κλάδο μας. Ε, το να φύγει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει να φύγει από την Ευρώπη. Αν ε, η Πρωθυπουργό Μέη το είπε αυτό και το εννοούσε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε ελευθερία, ελεύθερη κυκλοφορία των δημιουργών και των καλλιτεχνών πρέπει να διασφαλιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φρέζελ. Πάμε τώρα στην τελευταία μας εμπειρογνώμονα και αυτή θα μας παρουσιάσει τη Βρετανική πτυχή, τη Βρετανική οπτική. Η κυρία Έλουνετ Χαφ είναι η πρόεδρος του Wales Art International θα μας παρουσιάσει λιγάκι τον ε, οργανισμό της και μετά θα μας διαφωτίσει ε, σχετικά με το πώς θεωρεί η ίδια ότι το Brexit θα επηρεάσει τον ε, πολιτισμό και ε, τις δημιουργικές βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Είμαι η Πρόεδρος του Wales Art International μια, ε, ένας οργανισμός ε, του ε, Πολιτιστικού Συμβουλίου της Ουαλίας και με χρηματοδότηση από την Ουαλική κυβέρνηση. Θα επικεντρωθώ σήμερα σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Στους πολίτες και την ηθαγένεια, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την δημιουργική αλλά και τη γενικότερη οικονομία. Βέβαια, χρειάζεται κάποιο πλαίσιο πρώτα. Η Ουαλία είναι μία από τις τέσσερις περιοχές που αποτελούν τον το Βασίλειο στις δυτικές ακτές. Ε, μοιραζόμαστε την κελτική μας ε, πολιτική κληρονομιά με τα ε, κράτη της Ευρώπης και βεβαίως με ένα αμάλγαμα πολιτισμών στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το, η γλώσσα η ουαλική είναι γλώσσα μειονοτική και βεβαίως προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. η ταυτότητα είναι πραγματικά πολύ περίπλοκο θέμα και η διακυβερνητική δομή επίσης εξίσου δύσκολο. Η πολιτιστική πολιτική είναι ε, αποκεντρωμένο θέμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε υπάρχουν πάρα, πολλά, ε, πάρα πολλοί οργανισμοί που ασχολούνται με την εφαρμογή της. Το Brexit πραγματικά έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, οπότε είμαστε πολύ ευγνώμονες για τις πρωτοβουλίε που έχουν υπάρξει από το Βρετανικό Συμβούλιο και όλε τι υπόλοιπε φωνέ ε, σε Ευρώπη και ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τομεί μα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Οι ε, δημιουργικοί άνθρωποι ανθίζουν από, με, τις, με την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα όπω το Culture Action Europe, On the Move, το Literature Across Frontiers που ενώνει την Ευρώπη με του Βρετανού ομολόγου τη. Και πραγματικά πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργατική προσέγγιση. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο τομέας ε, δεσμεύεται σε ό,τι αφορά την ε, ε, διεθνή συνεργασία. 96% του τομέα ψήφισε υπέρ της παραμονής. ναι, όντως θα γίνει τώρα από το Brexit, αλλά πρέπει να, όταν θα ξανα διαπραγματευτούμε τις σχέσεις που θα δημιουργήσουμε, πρέπει να, είμαστε, να έχουμε τις σωστές συνθήκες για να προχωρήσουμε. Οπότε είμαστε όλοι ε, σε μια μεταβατική περίοδο. Ε, από το να παραμείνουμε πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές των πολιτιστικών τομέων της Ευρώπης που ε, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και, το, και προσπαθώντας να τους, να τους ξεχωρίσουμε είναι σαν να προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την ταπεισερή της Μπαγιέ. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε δουλέψουμε όλοι μαζί για την ειρήνη και την ευημερία. Mm. Όσο θα, όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ε, και τα διάφορα συμφέροντα διαγωνίζονται για την ε, προσοχή, δεν πρέπει να ξεχάσουμε Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον πολιτιστικό και ε, δημιουργικό κλάδο στην Ευρώπη. 87 ε, δισεκατομμύρια λίρες ε, προσθέθηκαν στο, στην, Ευρωπαϊ... Βρετανική οικονομία, 5,3% του το ΑΕΠ, 2 εκατομμύρια άτομα δηλαδή απασχολήθηκαν. 7% αύξηση από το 2014 και βεβαίω θα ήταν εύκολο η στραχτοπούτα να μην πάει στο χωρό παρόλο που είχε βάλει το φόρεμα για το χορό δεν, μπορώ, δεν θα σα μιλήσω βεβαίω μόνο για στατιστικά. Δεν είναι μόνο αριθμητικά στοιχεία τα σημαντικά, αλλά πρέπει να δούμε τι προσθέτει ο τομέα αυτό στην ποιότητα ζωή μα. Αυτό που έχουμε στην Ευρώπη είναι μια ενιαία αγορά του νου και βεβαίω αυτό το σεβόμαστε και, το, και μας είναι ιδιαίτερο πολύτιμο αυτό. Αυτή η φράση αναφέρθηκε από τον Γεράν Αλφάν Ντέιβις σε μια πρόσφατη έκθεση που έκανε για τον Brexit στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου λέμε ότι δεν υπάρχει μονοπόλιο ιδεών ή πολιτισμού, μπορεί, να, μπορεί να προκύψουν καλές ιδέες από μια ε, απομακρυσμένη περιοχή στη Δυτική Ουαλία ή από το Μπέρμιχαμ ή από το Λονδίνο ή από το Βερολίνο ή το Βουκουρέστι. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το οικονομικό κέρδος που δημιουργείται από την πώληση ενός πίνακα, για παράδειγμα. Ε, τέχνες τονίζουν πολλούς τομείς της ε, ζωής μας, από την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας, της, ε, την ε, επανακίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στα κέντρα των πόλεων, του πολιτιστικού τουρισμού δημιουργούν θέσεις εργασίας, εμπλουτίζουν τις κοινωνικές υπηρεσίες και έτσι φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Και έρχομαι στο πρώτο μου θέμα, τα άτομα και την ηθαγένεια η λίγο φράγκα των πολιτών είναι η συνεργασία. Αν δεν μπορούν να συνεργαστούν και δεν μπορούν να κινηθούν, σημαίνει ότι θα έχει αυτό τεράστιε συνέπειε και στον πολιτισμό και στην δημιουργική οικονομία τη Ευρώπη. Ήδη έχουμε ένα κενό σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε στην Ευρώπη και το να μπορούμε να έχουμε εργαζόμενου από πέρα των συνόρων μα είναι πάρα πολύ σημαντικό για του ε, τομεί αυτού. Και οι οργανώσει ε, τέχνη αλλά και οι επιχειρήσει έχουν τονίσει τι ε, αρνητικέ συνέπειε του Brexit. Τι μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε να βρούμε τρόπου για να διατηρήσουμε την ελευθερία τη διακίνηση των, των εργαζομένων αλλά και όλων των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι συζητήσει για τι ε, θεωρήσει ε, μικρή ε, διάρκεια μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τελικής συμφωνίας. Αλλά το πρώτο κομμάτι, το πρώτο βήμα είναι να δούμε το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι και αν γίνει, αυτός ο τομέα βασίζεται σε μια προσέγγιση συνεργατική οι εργαζόμενοι ε, πηγαίνουν εκεί που βρίσκεται η δουλειά. Ε, και το έχουμε δει και από ομάδες χορού, θεατρικές ομάδες, όπου υπάρχουν ε, πάρα πολλές ευκαιρίες να μετακινηθούν, αλλά με το Brexit δημιουργούνται πάρα πολλά προσκόμματα. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη ευαισθησία και οι ε, βαθιές σχέσεις που έχουμε με τα, ε, με τα Συμβούλια Τέχνης στην ε, Βόρεια Ορλανδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό περιβάλλον έτσι ώστε οι δύο οι, οι καλλιτεχνικές ομάδες να δουλέψουν απρόσκοπτα και στις δύο πλευρές. Δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον προσκόμματα. Ήδη υπάρχει οικονομική στενότητα, λιτότητα ε, και υπάρχουν πάρα πολύ, μεγάλοι, πάρα πολύ αυστηροί κανόνες ό,τι αφορά την κινητικότητα. Το δεύτερο είναι ο αντίκτυπο του Brexit στα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, στα προγράμματα που, χρησιμοποιούνται, που χρηματοδοτούνται συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Sage στο Gateshead, στο, στο Home του Manchester, από το Icon στο, του Birmingham μέχρι το Πόντιο στον Μπαγκόρ, τα προγράμματα που, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, βοηθήσει πάρα πολύ τα, τις πολιτιστικές υποδομές του Ηνωμένου Βασίλειου. Αλλά βεβαίως ε, ε, βλέπουμε ότι οι τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτές οι περιφέρειες να επηρεαστούν πάρα πολύ από την απόσυση αυτών των προγραμμάτων. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο όφελο στο να, να διατηρηθεί η συμμετοχή ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στα πολυμερή προγράμματα και για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω αυτό δεν είναι θέμα απλώ τη απώλεια ε, χρηματοδότηση. Τα δίκτυα και οι εταιρικέ σχέσει που έχει δημιουργήσει το Creative Europe ή οι υποδομέ που έχουν υπάρξει για τον τομέα μα, η εμπειρογνωμοσύνη είναι θέματα που δεν μπορούν να μετρηθούν με οικονομικούς όρους μόνο και ο αντίκτυπος της απόσυρσης αυτής της ε, χρηματοδότησης, ε, είτε είναι τα διαφορετικά ταμεία είτε το Creative Europe, δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με, συγκεκριμένες, ε, με χρηματοδότηση για συγκεκριμένα προγράμματα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που έχουν βραβευτεί ήταν, μάλιστα ήταν το Hinterland, ε, η απάντηση της ε, Ουαλίας στην, ε, στα φιλμ νουάρ των Σκανδιναβών. Παρήχθη στην Αγγλία, το είδαμε στο BBC και σε άλλα τοπικά κανάλια. Βρίσκεται σε πάνω, έχει πολιθεί σε πάνω από 30 χώρες και μπορείτε να το δείτε και στο Netflix. Ο Ed Thomas, ο, διευθυντής του, ο ε, σκηνοθέτης του Fiction Factory, ε, βλέπει πραγματικά τεράστια ωφέλη ε, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση από την Ευρώπη, όχι μόνο για την εταιρεία του και μάλιστα λέει ότι το να προωθούμε την πολυπικιλότητα του πολιτισμού και της γλώσσας στην Ευρώπη είναι σημαντικό και η εταιρική αυτή σχέση έχει δώσει φωνή σε μια μικρή χώρα στην, στον πολιτισμό της και στους ανθρώπους της. Η διατήρηση της, ε, του Creative Europe μαζί με τους άλλους ε, μη Ευρωπαίους εταίρους θα μας βοηθήσει να ε, δράσουμε και άμεσα και έμεσα. Σε ό,τι αφορά τον δημιουργικό τομέα, η συμμετοχή της του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πολλά ωφέλη. Αλλά δεδομένου ότι η, είναι αποκεντρωμένο καθήκον η, ο πολιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσαν τα κράτη της, του Ηνωμένου, που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο να, μην, να γίνουν μέλη μεμονωμένα του Creative Europe και να παραμείνουν εντό. Ο τρίτος τομέας είναι ο αντίκτυπος του Brexit στον, ε, στην ε, ε, δημιουργική και στην ευρύτερη οικονομία. Αν η ελευθερία της μετακίνησης των εργαζομένων είναι πραγματικά ο πυρήνας των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών, η πνευματική ιδιοκτησία είναι το νόμισμα του. Το Συμβούλιο της Αγγλίας ε, λέει ότι το δεύτερο, εξάμηνο, το δεύτερο τρίμηνο συγγνώμη, του 2016 78 εκατομμύρια τραγούδια και 51 εκατομμύρια ταινίε κατέβηκαν παράνομα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε είναι, είναι οι εταιρικέ σχέσει που μπορούν να μα υποφελήσουν αμοιβαίω. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν βασικέ βασικές ε, αρχέ ε, που θα τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και βεβαίω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον ορισμό των ευρωπαϊκών έργων. Υπάρχει ανάγκη και για το ΕΒ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν να συνεργάζονται ενεργά στην ψηφιακή ενιαία αγορά και κυρίω ό,τι αφορά την νομοθεσία για το copyright. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την δυνατότητα να ανταλλάσσουμε πληροφορίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, Ηνωμένου Βασιλείου χωρί να υπάρχουν περιορισμοί. Και τα δύο μέρη θα πρέπει να ε, σταματήσουν την, ε, να αντιταχθούν στην επιβολή δασμών στα πολιτιστικά, στα πολιτιστικά αγαθά και βεβαίω όλοι θα χάσουμε να σκοτώσουμε την κότα που πρόκειται να κάνει το χρυσό αυγό. Βεβαίω πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε δημόσια στήριξη για τα μέσα μαζική ενημέρωση και του δημιουργικού τομεί. Ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε την εξαίρεση της, ε, του πολιτισμού από τις ε, ευρωπαϊκές εμπορικές διαπραγματεύσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δημόσιες επενδύσεις γίνονται με διάφορους τρόπους για να βοηθήσουν τις δημιουργικές βιομηχανίες. Οπότε, όπως καταλήγω, θέλω να ζητήσω από εσά να ζητήσετε από τις εθνικές σας να στηρίξουν τη δημιουργική οικονομία και να συνεχίσουν την συνεργατική προσέγγιση με, πέραν του Brexit. Πρέπει να είμαστε παγκοσμιοποιημένοι, πρέπει να έχουμε όραμα για το μέλλον. Ε, γιατί η ευημερία της, και οι πολίτες της, ε, η ευημερία της Ευρώπης και οι πολίτες της Ευρώπης επηρεάζονται. Δεν πρέπει να ε, τους αστερίσουμε την ταυτότητα που έχουν θεωρήσει ως δεδομένη, αλλά να μην ε, εμποδίσουμε να είμαστε και ενεργοί ε, πολίτες, να μετακινούμεθα, να σπουδάζουμε σε άλλες ε, χώρες. Μην ε, έχετε αυταπάτες. Εγώ πιστεύω ότι το να δώσουμε στους πολίτες ένα μεγάλο φάσμα ε, διεθνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ουσιώδες για να έχουμε καλύτερες ε, σχέσεις που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό που υπάρχει τώρα παντού. Εγώ φοβάμαι για το μέλλον των παιδιών μου σε ό,τι αφορά τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν, τις πολιτιστικές, αλλά παραμένω αισιόδοξη ότι δεδομένων των αναλογιών και αν, υπάρξει, αν υπάρξουν ευκαιρίες, η επόμενη γενιά θα κάνει τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Ο τομέα για τον οποίο ενδιαφέρομαι τόσο πολύ ε, δίνει κάποιε ευκαιρίε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να υπάρξει καλύτερη κατανόηση που θα φτάσει πέρα από τα σύνορα. Ή ο πολιτισμό και η δημιουργικότητα έχει σημασία για όλου μα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε επιτυχεί. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, για τον ε, δημιουργικό κλάδο, για τον πολιτισμό. Έχουμε 13 λεπτά για τη συζήτηση. Και όπως ξέρετε πρέπει να ολοκληρώσουμε και στην ώρα μας. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στοργεύσκη και μετά στα υπόλοιπα μέλη που είναι εδώ, εφόσον το επιθυμούν. Παρακαλώ. Κοίτα, αναφερθήκατε εσείς ε, σωστά στα κυρίαρχα θέματα ας πούμε τις ε, εταιρείε οι οποίες ε, έχουν κάτω από 10 εργαζόμενους. Αυτοί ε, είναι που χρειάζονται και περισσότερη υποστήριξη γιατί αυτοί δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι γεγονός ότι οι καλλιτέχνες μετακινούνται για να συμμετάσχουν σε θεάματα, σε έργα κλπ. Κατά την δική μου άποψη, ε, η ευθύνη των διαπραγματεύσεων είναι μεγάλη ε, και βεβαίως θα πρέπει σε αυτές να εμπλακούν και ε, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες. Επίσης, εσείς αναφερθήκατε σε ποσοστώσεις, ποσοστώσεις συνολικές ή που να αφορούν μονάχα τους καλλιτέχνες. Επίσης, ε, τα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, μιλούν ε, για τον λόγο της, ε, της βασίλισσας ή περισσότερο ασχολούνται με το τι χρώμα είχε το καπέλο της παρά εάν, ας πούμε, είχε την ευρωπαϊκή σημαία κτλ. Κοιτάξτε, έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση της έντασης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο που όμως μειώνεται σιγά σιγά. Ναι, θα πρέπει να τη δω αυτή τη φωτογραφία, να δω τι καπέλο φορούσε και η Βασίλισσα. Ε, κρίμα, κρίμα που δεν είναι εδώ ο συνάδελφος ε, Φάρατς ε, του UKIP. Ε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εσείς στην ουσία, στην ουσία αυτό που προτείνετε απέναντι σε δύο μεγάλα ερωτήματα, ε, τον μεγάλο ρόλο που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, στην καλλιτεχνική παραγωγή και στο θέμα της ανακύκλωσης ας πούμε και μετακίνησης των καλλιτεχνημάτων, των έργων τέχνης κλπ και εσείς λέτε ε, ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ειδικό καθεστώς εάν ας πούμε παραμείνει ε, ε, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποια στρατηγική έτσι ώστε έτσι ώστε να αντικατα... αντισταθμίσουμε την έλλειψη και χρημάτων αλλά και διακίνησης καλλιτεχνικού προϊόντος. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δουλέψει πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα θέμα που είναι σημαντικό, το καθεστώς ε, του καλλιτέχνη. Ε, την επόμενη χρονιά είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά Πολιτιστικής Κληρονομιάς και δεν θα είναι ανοιχτή μονάχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως ελπίζω ότι θα αποτελέσει και μια καλή ευκαιρία ε, ανταλλαγής απόψεων για την πολιτιστική κληρονομιά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μιλάμε για πολύ λίγα άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Έχει υποθεί πολλές φορές στη συζήτηση ότι αυτά τα ζητήματα που εξετού, εξετάζουμε όσον αφορά τον πολιτιστικό και το δημιουργικό τομέα, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και βεβαίως η ενιαία αγορά είναι ζωτική σημασίας και για τις θέσεις εργασίας ε, για τις οποίες επίσης μιλούμε πολύ, έχω την εντύπωση ότι μιλάμε σε μια γλώσσα που ο κόσμος κανονικά, που συνήθως δεν καταλαβαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μιλάμε για τον τομέα ε, του πολιτισμού και το δημιουργικό τομέα, ενώ μιλάμε για κάτι το οποίο συναισθηματικά αφορά πολύ τον κόσμο και είναι πολύ κοντά στον κόσμο. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορούμε να το περάσουμε αυτό, ειδικότερα στους νεότερους που πηγαίνουν σε φεστιβάλ μουσικής, ε, που συμμετέχουν σε συγκροτήματα, που ταξιδεύουν στο εξωτερικό κλπ να του εξηγήσουμε ενδεχομένω ποιο θα είναι ο αντίκτυπο αυτή τη κατάσταση για ένα θέμα που ε, του απασχολεί πάρα πολύ και του ενδιαφέρει πολύ ότι αυτό ο τομέα ναι, μεν δημιουργεί θέσει εργασία, αλλά πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένας καθημερινός αντίκτυπος όλων αυτών των ε, αλλαγών που ενδεχομένως ε, θα ε, συμβούν και ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε για να το επιτύχουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο τώρα στους ε, δύο εμπειρογνώμονές μας. Όποιος θέλει να ξεκινήσει μπορεί να ξεκινήσει. Um, Εγώ θα ξεκινήσω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα θέματα. Ε, ίσως να ξεκινήσω από το τέλος. Καθημερινή ζωή, καθημερινή εμπειρία της καθημερινής ζωής. Ε, είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, ε, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, δεν έχει γίνει συζήτηση, ε, εθνική συζήτηση για τον αντίκτυπο που θα έχει ε, το Brexit στο... θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει όμως μια τέτοια συζήτηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επομένως οδηγούμε και στο ερώτημα γιατί στην Ευρώπη των 27 ε, γιατί τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες και οι καλλιτέχνες δεν υψώνουν το ανάστημά τους για να πούν είμαστε αντίθετοι στο Brexit και να κλείσουν μια μέρα ας πούμε και τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες και τα λοιπά. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ε, και ο τομέας ε, της, ε, του πολιτισμού θα πρέπει απέναντι στο Brexit να αναλάβει τις ευθύνες του και να δει και πόσο αντίκτυπο έχει στον κόσμο. Ναι, βεβαίω οι κυβερνήσει, ε, εγώ λέω και όχι και σε σχέση με την άλλη ερώτηση, ε, οι κυβερνήσει και όχι οι ε, οργανώσει κλπ. θα έχουν την ευθύνη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει έρθει όμω κανένα σε επαφή μαζί μας για να δουν ποια είναι η άποψη της βιομηχανία, τη δημιουργία της για το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το ειδικό καθεστώς, ε, το ανέφερε η κυρία Κώστα αυτό. Νομίζω ότι ε, το θέμα της εξαίρεσης ε, του πολιτισμού είναι κάτι που και οι δύο πλευρές θέλουν. Και νομίζω ότι το νορβηγικό μοντέλο είναι το πιο κοντινό. Το σημαντικό είναι να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, με τρόπο ώστε ε, να γίνει κατανοητό ότι ε, θα χρειάζεται πενταετής αναθεώρηση της ε, μετα-Brexit περίοδου έτσι ώστε να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Δηλαδή το σημείο της αποχώρησης, το σημείο, η χρονική στιγμή του Brexit δεν θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο ολοκλήρωσης αλλά περισσότερο ένα σημείο εκκίνησης. Θα πρέπει μάλιστα στο τομέα του πολιτισμού για να θεωρήσεις να γίνουν και πιο κοντινά, δηλαδή κάθε δύο, κάθε τρία χρόνια και όχι κάθε πέντε ή δέκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χάφ. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω και ο πολιτισμός είναι οπωσδήποτε άρρηκτα συνδεμένος με όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μάλλον ε, πολύ σημαντικό συστατικό κομμάτι. Χρειαζόμαστε επαφές, χρειαζόμαστε να συνεχίσει η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δούμε βεβαίως και την ίδια τη δομή των διαπραγματεύσεων ε, και είναι αλήθεια ότι δεν ακούγεται πάντα σε ικανοποιητικό βαθμό η φωνή του πολιτισμού. Δεν, γιατί είναι πολυσχηδής ο πολιτισμός και εκφράζεται με πάνω από μία φορά. Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά του πολιτισμού και της ε, ε, βιομηχανίας, ε, της ψυχαγωγίας, της παραγωγής, της δημιουργίας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με τα μέλη μας και να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Αλλά μια και αναφέρθηκε μάλιστα και το Βρετανικό Συμβούλιο, το British Council, είναι σημαντικό να μιλούμε με τους εταίρους μας για να μιλήσουν και εκείνοι να ακουστεί η φωνή τους στις δικές τους κυβερνήσεις και οπωσδήποτε σε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε σημείο καταλήξουμε θα πρέπει να έχουμε καταλήξει όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Äh, äh, Βεβαίω. Μπορείτε να απαντήσετε ε, αν θέλετε, αλλά πολύ σύντομα. Δεν έχουμε απαντήσει στις ε, ρωτήσεις των ε, φοιτητών από το Μάντσεστερ. Το σημαντικό είναι να ξέρετε ότι παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξακολουθήσετε να είσαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της κοινότητας των Ευρωπαίων. Οπότε μάθετε γλώσσες, ταξιδέψτε, φέρτε ε, τη δική σα κουλτούρα στην υπηρετική Ευρώπη. Εμένα πάντα μου άρεσε το, όταν ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε να είστε κομμάτι της Ευρώπης παρόλο που δεν θα είστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ενθαρρυντικά τελευταία σχόλια για τους ε, προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ε, κυρίως τους εμπειρογνώμονές μας οι οποίοι νομίζω ότι μας έδωσαν πολλές, πολλά ενάβσματα για τις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε βέβαια στην αρχή ακόμη και η Επιτροπή Πολιτισμού και εκπαίδευση θα εμπλακεί ενεργά σε όλη τη διαδικασία που έχουμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Σίγουρα θα μας ζητηθεί ε, Ο Γκίφερ Χόφστατ ούτω ή άλλω θα είναι στι διαπραγματεύσει. Θα μα ζητηθεί λοιπόν να δώσουμε και εμεί τη γνωμοδότησή μα για το ένα ή το άλλο θέμα, για τα θέματα τη εκπαίδευση, του πολιτισμού. Και νομίζω ότι σήμερα πραγματικά ακούσαμε πολύ σημαντικά θέματα, μάθαμε πολλά και Τώρα ποιο θα είναι ο, ο, ο συνομιλητή μα στο Brexit για, τον πολιτισμό και τις, ε, Δημιουργικέ βιομηχανίε. Ο κύριο ε, Μπαρνιέ θα το κανονίσει αυτό. Αλλά βεβαίω η Επιτροπή Πολιτισμού θα είναι η καθήλυνα αρμόδια για όλα αυτά τα προγράμματα και για όλα όσα απορρέουν από αυτά τα προγράμματα. κλείνοντα να πω ότι ο πολιτισμό και η εκπαίδευση είναι μεγάλο κομμάτι που έχουν, που, και έχουν να κάνουν με, την, ε, με το να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, είτε είναι στην δημιουργική βιομηχανία, είτε στον πολιτισμό, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης, των, ε, της εργασίας των νέων και νομίζω ότι ως προς αυτό θα παρακολουθήσουμε όλοι τις ε, ε, διαπραγματεύσεις, όχι να διαλέγουμε και να παίρνουμε ό,τι μας συμφέρει, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να συνδέσουμε τους ε, ανθρώπους που βρίσκονται από την αποκή της μάχης. Αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ όλους, καλό σας απόγευμα και πάλι ευχαριστώ τους ε, παρασκεκλημένους μας. Και βεβαίως πέρα στις συνεδρίασεις. Και η πρόεδρος ευχαριστεί και τους δερμηνείς και εμείς την ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.